Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το νίκο της δημοκρατίας. Το μόνο θεσμικό όργανο που εκλέγεται το μόνο θεσμικό όργανο, ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που εκλέγεται από τους πολίτες. Σας εύχομαι το καλώς ήρθατε. Κάθε βουλευτής εκπροσωπεί τους συμπολίτε του. Καλώς ήρθατε όλοι. Καλή δουλειά εύχομαι στους νέους, στους νέους ευρωβουλευτές. Καλημέρα σε όλους. Δυνάμει του άρθρου της 20 Σεπτεμβρίου του 1976 που αφορά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την πράξη αυτή με καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 154 παράγραφος 2 του κανονισμού του Κοινοβουλίου κηρύσσω την έναρξη της πρώτης συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα Λοιπόν, θα ακούσουμε τον ύμνο της Ναέσκανος και σηκωθούμε να ακούσουμε τον ύμνο τον Ευρωπαϊκό. Είναι θέμα σεβασμού να σταθούμε όρθιοι. Δεν έχει σχέση με το αν συμμεριζόμαστε την άποψη του Όταν ακούμε τον ύμνο μια χώρα, σηκωνόμαστε όρθιοι κανονικά. Προσοχή. Να υπενθυμίσω ότι μην το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού του Κοινοβουλίου υπό την Προεδρία του βουλευτού που προσωρινά εκτελεί καθήκοντα Προέδρου δεν μπορεί να λάβει χώρα καμία συζήτηση της οποίας αντικείμενο να είναι εκτός του θέματος εκλογής του Προέδρου ή της ε, παλήθευσης εξακρίβησης των εξουσιών. Εγώ προεδρεύω αυτή τη συνεδριάσεως όπως το βλέπει ο κανονισμός, ότι ο απερχόμενος πρόεδρος ε, είναι εκείνος που ε, προεδρεύει προσωρινά στην Σύνοδο του Κοινοβουλίου. Όλα τα επίσημα έγγραφα που αποτελούν τη βάση για την εκλογή των βουλευτών θα διαβιβαστούν στην αρμόδια επιτροπή για την επαλήθευση των εξουσιών και θα δημιουργηθεί δυνάμει του άρθρου 206 του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ε, όσο οι εξουσίες ενός βουλευτού δεν έχουν επαληθευτεί ή αν δεν έχει αποφασιστεί επί τους ουσίας ελεγχόμενη ένσταση ο βουλευτής έχει πλήρη δικαιώματα στο Κοινοβουλίο και στα όργανα του Κοινοβουλίου από τη στιγμή που έχει υπογράψει την γραπτή δήλωση ε, μη ασυμβατότητας οι βουλευτές που καλύπτουν μια θέση που είναι ασύμβατη με αυτή του βουλευτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ταινία του άρθρου 7 της πράξεως της 20 Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, άμεση ψηφοφορία, δεν δίνονται να ε, καταλάβουν το αξίωμά του τη θέση τους. Για να μπορέσουν να απολαύσουν των πλήρων δικαιωμάτων των 29 βουλευτέ που δεν έχουν ακόμα υπογράψει την δήλωση μία συμβατότητα, καλούνται να το κάνουν αμέσω. Στι θέσει εκεί που βρίσκονται στην έσω κυκλίου. εκεί που βρίσκονται τα έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση, αύριο δεν θα έχουν την έγκριση, την δυνατότητα, την εξουσία να ψηφίσουν. Αύριο το πρωί θα προβούμε στην εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού μας κανονισμού. Δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 οι υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου του Κοινοβουλίου θα πρέπει να υποβληθούν με τη συνένεση των υποψηφίων από μια πολιτική ομάδα ή από τουλάχιστον 38 βουλευτές. Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιωτήτων εκπνέει σήμερα στις 22, ώρα 22. Λοιπόν, τώρα Πάμε στην κλήρωση για τον διορισμό των οκτώ ε, ψηφολεκτών. Θέλετε να μιλήσετε για την ψηφοφορία και μόνο. Δεν Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε το λόγο για την εκλογή του Προέδρου. Δεν μπορείτε να μιλήσετε μόνο για την εκλογή του Προέδρου αν θέλετε κάτι για τη διαδικασία σε ό,τι αφορά τους κανόνες που αναφέρατε και τις, ε, την εντολή των βουλευτών, θέλω να συγχαρώ όλους τους βουλευτές που εξελέγησαν και βρίσκονται εδώ σήμερα. Δυστυχώς όμως ορισμένοι βουλευτές που έχουν εκλεγεί δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την αίθουσα. Τρεις εκπρόσωποι του καταλανικού λαού δεν έχουν ε, το δικαίωμα πρόσβασης. Τους αρνήθηκαν το δικαίωμα πρόσβασης. Ε, Αυτό είναι ο οίκος της δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς που εκπροσωπούμε τα δικαιώματα και του λαού της Καταλωνίας ε, πρέπει να τα σεβαστούμε, αλλιώς τίθεται η αμφισβήτηση και η αξιοπιστία ε, του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει εκ μέρους των εκλεγέντων βουλευτών να κάνετε μια δήλωση κύριε Πρόεδρε για να επανεπιβεβαιώσετε την ισχύ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξία τους. Πάμε λοιπόν στην κλήρωση για, την, ε, τον διορισμό, τον καθορισμό των οκτώ ψηφολεκτών. Συνάδελφος Γιάν Όλμπερτ, δέχεστε να παίξετε το ρόλο του ψηφολέκτου. Πέτερ Πέτερ Γιάρ, δέχεστε ε, το ρόλο του ψηφολέκτη. Συνάδελφε Ένικ Όβερκαρντ Νίλσεντ, δέχεστε να είστε ψυχοφολέκτης. Συνάδελφε Γέρζι Μπούζεκ, δέχεστε να είστε ψηφολέκτης. Θα έχουμε έναν πρώην πρόεδρο ψηφολέκτη. Πολύ έμπειρος. Μπερνάρ Γκουέτα, δέχεστε να είστε ψηφολέκτης. Είστε παρόν, έτσι. Αλεξάνδρα Λέσλι Φίλιπς, δέχεστε να είστε ψηφολέκτρια. Ε, κοιτάξτε, δεν, δεν, δεν κάνετε τον υποστηριχτή, το φίλο άνθρωπο τη ομάδα. Μπάρμπαρα Τάλερ, δέχεστε να είστε ψηφολέκτης. Eh. Είναι παρούσα. Είναι παρόν. Όχι. Συνάδελφε Κατρίν Σαμπό, δέχεστε τη θέση του ψυχολέκτη έχουμε ψηφολέκτες τους εξής. Olbricht per, onorevole, per l'urna AB. Onorevole per l'urna CD. Για την CD, κύριος Γιάρ. Overguard για την για A μέχρι G τα ονόματα. Κύριος Μπούζεκ από Α, από Ι μέχρι Γκουέτα. Γκουέτα από LM, λάμδα μη. Τάλερ για την κάλπη N μέχρι ρο, Σαμπό S μέχρι ταφ, Φίλιπς. από U μέχρι ΖΙΤΑ. Παρακαλούμε τους ψηφολέκτες ε, να έρθουν στο, εδώ, στη θέση του Πρόεδρου. Η εκλογή του Πρόεδρου θα λάβει χώρα αύριο στις 9 το πρωί. Λοιπόν, διακόπτη συνεδρίαση.